Buongiorno colleghe e Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως μπορείτε να καθίσετε για να ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες. L'ordine del giorno θα ψηφίσουμε λοιπόν για την ε, έκθεση του κυρίου Γκιόνις ε, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Πρόκειται για μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Οι ε, τροπολογίες από το 35 έως το 44 απεσύρθησαν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε για ε, το ε, ένα συμβασμή υπέρ, κατά, αποχές, ο, το μπλοκ υπερθμών ένα συμβασμός εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών 11 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 533 υπέρ, 67 υπέρ, 453 κατά. Η τροπολογία αριθμών 11 απορρίπτεται. Έτοιμα ονομαστικής ψηφορίας για το 13. Αυτή αποσύρεται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, συνάδελφε. Πρόεδρε, δεν λειτουργεί ε, το δικό μου το μηχάνημα και στην ε, προηγούμενη ψηφορία υπερψήφισε, αλλά δεν λειτουργήσε το ε, μηχάνημα που έχω μπροστά μου. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα στείλουμε πάρα αυτά έναν τεχνικό για να επισκευάσει την, το μηχάνημα της ψηφοφορίας μπροστά σας. Περνάμε στο 14 μονομαστική ψηφορία. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 566 παρόντες, 94 υπέρ, 351 κατά. Η τροπολογία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 51 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 570 παρόντες, 488 υπέρ, 80 κατά, ε, δύο εποχές. Η τροπολογία υπαριθμών 51 εγκρίνεται. Τροπολογία 1 και 45 ως εκ τούτου καταπίπτουν. Ψηφίζουμε για τις ε, τροπολογίες 15 ε, και 46 με ονομαστική ψηφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε η ψηφοφορία. παρόντες 578, ε, 73 υπέρ, 491 κατά ή ε, οι τροπολογίες 15 και 46 απορρίπτονται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 65 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. παρόντες 587, 492 υπέρ, 81 ε, κατά. Η τροπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για τις τροπολογίες 67-68 από κοινού. Ψηφίζουμε για αυτές τις δύο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Εγκρίνονται οι τροπολογίες. Ψηφίζουμε για την 18 και 50 που είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Παρόντες 594 υπέρ 70, 522 κατά ως εκ τούτου οι τροπολογίες απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα για την 69, ε, την τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές η τροπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 21 και 47 ταυτόσημες ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Παρόντες 596, 89 υπέρ, 372 κατά. Οι ε, τροπολογίες απορρίπτονται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 48 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Παρόντες 602. Υπέρ 72. Κατά 518. Η τροπολογία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία υπερθυμών 49 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Παρόντες 605, ε, 86 υπέρ, 518 κατά. Η ε, τροπολογία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 82 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 54 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ως εκ τούτου η τροπολογία υπαριθμών 4 καταπίπτει. Ψηφίζουμε για την 5 την τροπολογία μονομιστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Η ψηφοφορία έκλεισε. Παρόντες 609 υπέρ 90, 383 ε, κατά η τροπολογία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 56 ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Η... Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Παρόντες 608, 516 υπέρ, 66 κατά. Η τροπολογία εγκρίνεται. Για την 81 ψηφίζουμε την τροπολογία, ε, η οποία αποσύρθηκε, με συγχωρείτε. Ως εκ τούτου ψηφίζουμε για την 55, για την τροπολογία 55. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές η τροπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την πρόταση της Επιτροπής ε, ως τροποποιήθηκε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές η πρόταση εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Παρόντες 602, 516 υπέρ, 82 κατά. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Ντόνσ. Τώρα περνάμε στις ε, δηλώσεις ψήφου επεξηγής ψήφου, με συγχωρείτε, επεξηγής ψήφου. Και δίνω το λόγο στον κύριο Άλντο Πατρίτσέλο για ένα λεπτό.